περίοδο Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται. Εύχομαι σε όλους τους αδέλφους ασφαλή επιστροφή και αναζωογονητικές θερινές διακοπές. Με χαρά να σας ξαναδώ το φθινόπωρο φρέσκους και ξεκούραστους.